hello Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση αυτή της Οικονομικής Επιτροπής. Τη μισή ώρα που καθυστερήσαμε ελπίζω να την χρησιμοποίησατε με χρήσιμο τρόπο. Είναι το θέμα του προϋπολογισμού που αναβλήθηκε και το κύριο Γκάλερ είχε μια πρόβλεπτη συνάντηση των συντονιστών όπου ήταν αναγκαίος. Γι' αυτό και δεν ε, θα είναι εδώ. Ε, έγκριση ημερήσιας διάταξης. Παρατηρήσεις. Όχι, εγκρίνεται. Και έχω μία μικρή ανακοίνωση. Προσοχή. Σας ενημερώνουμε ότι αύριο το πρωί, επειδή θα έχουμε κοινή συνεδρίαση με τους προπολογισμού για την Ευρωζώνη, θα καθαριστεί η αίθουσα, θα ξαναφτιαχτεί για αύριο το πρωί και θα καθόσαστε αλλού από όπου κάθεστε τώρα. Δεν ξέρω με τι κριτήρια, αν θα χωριστούμε προπολογισμοί οικονομικοί, πάντως οι υπηρεσίες θα αναδιατάξουν την αίθουσα. Οπότε να πάρετε τα πράγματά σας μαζί σας σήμερα το βράδυ, γιατί αύριο θα κάθεστε κάπου αλλού. Και ερχόμαστε έτσι στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Πράσινη βίβλος για αλλιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Λότριξον, έχεις το λόγο. Παρακαλώ. Ε, vi inleder idag ett mycket intressant arbete.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 Εμεί ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά, λέει ο Πρόεδρο. και τώρα ισχυώδης εισηγητής πρώτα απ' για το Λεκό Κόμμα, τον Αντικαντελάρ. Τον κύριο Καντέκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε σήμερα, είπε ο σχεδόν συγχητή και θέλει να πω ότι εδώ και 8 χρόνια και περισσότερο έχουμε την πρώτη πράσινη εκδοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά τι χρηματοδομικέ υπηρεσίε και δημοσιοποιήθηκε. Όμω θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι αυτέ οι υπηρεσίε ακόμα είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένε σε εθνικό επίπεδο και όλα αυτά έχουν επιτευχθεί κάποια πράγματα. Πρώτα-πρώτα εγκρίναμε πάρα πολλά κείμενα τα οποία θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα των καταναλωτών σε αυτά τα ε, αξιόγραφα ελληνική. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να γίνει μεταφορά στο εθνικό ε, δίκαιο. Και επίση θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η η νομοθεσία πριν νομοθετήσουμε εκ νέου. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκροτήσει μια ψηφιακή αγορά και μια κεφάλαιο αγορά, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε μια αυθεντική αγορά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής επίση, Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με κάποια προβλήματα για τις υπηρεσίε για αυτές τις, ε, τις αλλαγές οπότε θα πρέπει να δούμε ότι ο ανταγωνισμός φέρνει κάποια θετικά πρώτα πρώτα οθεί στην καινοτομία έτσι αυξάνονται οι επιλογές αλλά και η ποικιλία των προϊόντων ε, και κατεβαίνουν οι τιμές ε, υπέρ του καταναλωτή ε, οπότε όσον αφορά τις αλλαγές λιανικής έχουμε τα προβλήματα Υπάρχει η τραπεζική παράδοση των κρατών μελών, υπάρχει το θέμα της γλώσσας αλλά και της εμπιστευτικότητα. Και ο καταναλωτή αυτών των υπηρεσιών θα ε, απευθυνθεί σε κάποια εταιρεία κοντά του και θα επικοινωνήσει με εκείνη, θα ζητήσει συμβουλές στη γλώσσα του. Και θα πρέπει να την εμπιστεύεται. Ακριβώ το ίδιο ισχύει και για τι τράπεζε. Οι τράπεζε δυσκολεύονται τα, να προωθήσουν τα προϊόντα του ε, στο εξωτερικό. Γιατί εκεί το περιβάλλον και το νομοθετικό αλλά και η ε, τραπεζική παράδοση διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Οπότε η πραγματική πρόκληση είναι ότι θα πρέπει να δημιουργούν κάποια κίνητρα για αυτέ τι ε, δραστηριότητε, τι διασυνοριακέ και από πλευρά προσφορά αλλά και ζήτηση. Η δε ψηφιοποίηση είναι το μέσο για να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι, αλλά δεν αρκεί. Γιατί ε, οι δυνατότητές μας παραμένουν περιορισμένες. Να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Θέλουμε να υπάρχει μια αγορά. Ε, το πενευόμαστε, αλλά όμως από την άλλη μεριά, τα ε, δικαιώματα των, καταναλωτών και όλες οι σχετικές ρυθμίσεις ανήκουν στο εθνικό επίπεδο. Οπότε έχουμε μια αγορά, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε 28 ε, διαφορετικά καφρολογικά δίκαια οπότε θα πρέπει τώρα να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε την υπόθεση αυτή για τα ΜΜΕ και όλα τα κρατημέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα νομοθετικό οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον το οποίο είναι προσυρμοσμένο στι ιδιοτυπίε των ΜΜΕ γιατί είναι η ΜΜΕ η σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας δημιουργούν απασχόληση αλλά και ανάπτυξη θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβασή του στην χρηματοδότηση αυτό να είναι θέμα προτεραιότητο. και από αυτή τη πλευρά θα πρέπει οι τράπεζες να ε, δανείζουν στις ΜΜΕ και θα πρέπει οι ευκολίες αυτές να αυξηθούν. Οπότε οι καταναλώτες επίσης θα πρέπει να εμπιστεύονται τα προϊόντα και αυτούς που παρέχουν τα προϊόντα. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι στις ανάγκες τους. Αλλά χρειάζεται ε, πλήρης ενημέρωση. Ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να έχει προστασία ε, και στον δικαιώματά του παντού στην Ευρώπη κατά τον ίδιο τρόπο. Και αυτό θα πρέπει να κατοχυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη οι δε πάροχη των χρηματοοικονομικών προϊόντων ε, λιανικής και των σχετικών προϊόντων θα πρέπει να παράσχουν εγγύσεις προς τους πελάτες τους και να δίνουν τις σημαντικότερες πληροφορίες και έτσι να μπορεί ο πελάτης να αναπτύξει δυνατότητες καινοτομίας και θα πρέπει όλοι επομένω να έχουν τα κατάλληλα κίνητρα για να δημιουργήσουν κάποια τραπεζικά προϊόντα προσβάσιμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις ιδιοτυπίες του καθενός των εμπλεκομένων και τις ιδιοτυπίες του κάθε προϊόντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει κάποιες προτάσεις που οπωσδήποτε θα βοηθήσουν να αναπτυχθεί προβληματική για τις ε, διασυνοριακές ε, ε, συναλλαγές και για το πώς θα υπάρξουν κάποια πανευρωπαϊκά προϊόντα σε αυτόν τον τομέα. Και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, ECR. Ashley Fox. Ή εκ μέρους του Ashley Fox μάλλον. Ευχαριστώ αντιπροσωπώ τους περισσότερους ε, συναδέλφους σήμερα, οπότε θα ξαναπάρω τον λόγο. Ο Ασλή ζητάει τον λόγο, καλωσορίζει την προσέγγιση της Κομισιόν ιδιαίτερα την ε, θέση ότι πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου πριν προχωρήσουμε σε παραπέρα νομοθεσία. Είναι σαφέ βεβαίω πως δεν υπάρχει μια σαφή ενιαία εσωτερική αγορά για τι υπηρεσίε αυτέ. Ε, το επίπεδο διασυνοριακών συναλλαγών είναι μόνο 1% και θεωρεί πως υπάρχουν κάποια φυσικά εμπόδια που ε, αναγκάζουν του καταναλωτέ να επιλέγουν τοπικού παρόχους. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έτσι θα μπορούσαν να αναλάβουν οι πάροχοι μεγαλύτερο κίνδυνο και να, να ανέβει το κόστος σε κάποιε χώρε. Μία ανησυχία που έχει ο συνάδελφο είναι το κατά πόσον θα εφαρμοστούν κάποια τέτοια μέτρα στην πράξη. Από τη σκοπιά της ασφάλιση, ε, τα διαφορετικά νομικά συστήματα θα μειώσουν τη δυνατότητα μεταφορά των ε, συμβάσεων αυτών διασυνοριακό. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην αυξανόμενη διασυνοριακή δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε, όπω παραδείγματο χάρη η αύξηση των καταναλωτών στι λιανικές χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και η ενίσχυση του ανταγωνισμού. Το θέμα της εμπιστοσύνης ε, των καταναλωτών ε, μέσω ακριβέστερων πληροφοριών για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές των υποπτικών αρχών θα επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα και έτσι θα μπορούσουμε μέσω και του συστήματος εγγύησης καταθέσεων να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο κάλυψης σε ολόκληρη την Ένωση. Όσον αφορά την προώθηση του ανταγωνισμού πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα βλέπει αυτές τις εταιρείε ως εταιρείε οι οποίες δημιουργούν ευκαιρία και όχι μόνο κίνδυνο. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να γίνουμε μια παγκοσμίω πρωτοπόρος ε, αγορά και υπάρχει επίσης ε, στις είπα και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το οποίο λέμε το ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο δοκιμάζονται κάποια πράγματα όπως το crowdfunding το οποίο δίνει μεγάλες δυνατότητες μάλιστα μία παρατήρηση του Προέδρου για το Περιπάνω των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κυρία Νετφέλτ, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή που δήλωσε πως θέλει να βρεθεί συνένεση με όλες τις ομάδες και καλωσορίζω και τις δηλώσεις των άλλων συναδέλφων, ειδικά του ΕΛΚ που λέει πως ε, υπάρχει ένα επίπεδο φιλοδοξίας και νομίζω πως αυτό είναι βασικό γιατί στο τωρινό πολιτικό κλίμα έχουμε σημειώσει εδώ και αρκετά χρόνια πως ακόμα και οι πιο ευρωσκεπτικιστές ε, είναι υπέρ της εσωτερικής αγοράς, αλλά στην πραγματικότητα λίγα συμβαίνουν και έχουμε δει κάποια σχετικά θέματα όπως τις οδηγίες ΜΥΦ των ενδιάμεσων ασφαλιστών όπου προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια εσωτερική αγορά και βλέπουμε ότι στην πράξη τα κράτη-μέλη μπλοκάρουν οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο και θεωρώ πως τα κράτη-μέλη πρέπει να ρωτηθούν εάν ε, παίρνουν στα σοβαρά την ενιαία αγορά ή αν προτιμούν να συνεχίζουν να μιλούν για εθνική κυριαρχία. Γιατί αν ισχύει αυτό δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ενιαία αγορά. Αν θέλουμε να έχουμε ενιαία αγορά δεν πρέπει να υπάρχουν ταμπού. Οι φορολογικές πτυχές δεν πρέπει να είναι ταμπού. Η διασυνοριακή προστασία των καταναλωτών και εναρμόνιση επίσης και η μεγαλύτερη εναρμόνιση δεν θα πρέπει να είναι ταμπού. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απαντήσουν το ερώτημα αν έχουν την πολιτική βούληση για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Γιατί βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι εθνικές πρακτικές. Μπορούν αυτό να το πούν στους ψηφοφόρους τους. Αναφέρθηκε ήδη η λέξη χρηματοπιστωτική τεχνολογία και κοιτάξτε, αν συνεχίσουμε να διστάζουμε θα μας ξεπεράσει η πραγματικότητα. Η τεχνολογία θα βρει τον τρόπο της, θα διαταράξει τα συστήματα και αν δεν έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει αλλού οι μεγάλες εταιρείες ήδη λένε πως θα φύγουν από την Ευρώπη γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φραγμοί εδώ πέρα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε φιλοδοξία, να είναι η Ευρώπη η έδρα της τεχνολογίας της ε, χρηματοπιστωτικής ή όχι. Ή θα κάνουμε ό,τι κάναμε σε άλλα πράγματα, θα μιλάμε δηλαδή επί χρόνια και με πενιχρά αποτελέσματα. Γιατί ειλικρινά σα λέω, έχουμε και δουλειέ. Έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε, αν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ταμπού και εδώ πέρα θα ήθελα να πάω ακόμη και παραπέρα και από τον συνάδελφο του Λαϊκού Κόμματο που λέει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι δεδομένα η εθνική κυριαρχία και οι αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας. Ναι, ταυτόχρονα Έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες της Ευρώπης που περιμένουν κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Οπότε πρέπει να είναι φιλόδοξη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει κάποια πραγματική προοπτική στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Σόφη. Δεν βλέπω κάποιον από την ΚΟΕ. Περνάμε λοιπόν κατευθείαν στους πράσινους. Σβέν Γκίγκολντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα ακούστηκαν. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τα ξεκάθαρα λόγια του για μια προσέγγιση με βάση τη συνεργασία οπωσδήποτε. Εμείς ως πράσινοι καλωσορίζουμε την πράσινη βίβλο και βλέπουμε πως ε, το Κοινοβούλιο πραγματικά επιδεικνύει μια φιλοδοξία και ότι δεν έχουμε απλά έναν κατάλογο θεμάτων εδώ πέρα. Πιέζουμε κοινοβούλιο, ε, Συμβουλίο και Κομισιόν να φέρουν μέτρα τα οποία θα υλοποιήσουν την φιλοδοξία αυτή. Από τη δικιά μας σκοπιά τώρα υπάρχουν κάποια ζητήματα υπάρχουν καταναλωτές ε, και επενδυτές οι οποίοι υποφέρουν ε, από την επιθετική τιμολόγηση και δεν ε, αμείβονται αρκετά για το ρίσκο το οποίο αναλαμβάνουν και πολλοί καταναλωτές και επενδυτές δεν λαμβάνουν τις αποδόσεις που θα έπρεπε να έχουν. Πολλά λεφτά σπαταλούνται σε ένα σύστημα ενδιαμέσων το οποίο είναι υπερτροφικό. Και ο σκληρότερος ανταγωνισμός και το άνοιγμα των συνόρων μπορεί ακριβώς να μειώσει αυτά τα φαινόμενα. Οπότε η βασική προσέγγιση νομίζω ότι της Κομισιόν είναι καλοδεχόμενη για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο περισσότερων αποδόσεων για τους επενδυτές πρέπει να τυποποιήσουμε τα προϊόντα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες για να υπάρξει αποτελεσματικός ανταγωνισμός και άρα να προσφέρουμε απλά και ασφαλή και φτηνά προϊόντα. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν απλούστερα και καλύτερα συστήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει ακριβώς ο ανταγωνισμός και η διασυνοριακή σύγκριση. Και εδώ πέρα έχει μεγάλη σημασία να φροντίσουμε η τροπολογία αυτή να είναι μόνο μία από τις δυνατότητες διασυνοριακής τυποποίησης. Τέλος, οφείλω να πω πως δυστυχώς, και εδώ πέρα θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Κομισιόν το η πράσινη βίβλος δεν ήταν πράσινη. Δηλαδή, πολλοί επενδυτές θέλουν να κάνουν την διαφορά με τις επενδύσεις τους, να βοηθήσουν να επιτευχθούν οι στόχοι της διάσκεψης του κλίματος. Αλλά να υπάρχει και ένα αηφόρο γενικότερα περιβάλλον. Αλλά δυστυχώς στην Πράσινη Βιβλία δεν έχετε τίποτα το ουσιαστικό προς αυτή την ε, κατεύθυνση για να βοηθήσετε ακριβώς ε, το πράσινο αυτό θέμα. Και ειδικά όσον αφορά θέμα και θα έπρεπε ακριβώ να προωθήσετε την πράσινη και αηφόρο, τις αηφόρες κρηματοοικονομικές λύσεις. Εμείς ευχαριστούμε Σβέν και τώρα ο σκιώδος του EFDD. Παρακολουθείς το λόγο. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Δεν έχω να επικνούν ιδιαίτερα στο κείμενο αυτό. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε σε μια πλατφόρμα πέντε βασικών αργών. Βέβαια θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια στην ε, ενημέρωση ε, για όλους όσους θέλουν να επενδύσουν, δηλαδή να έχουν επίγνωση του τι κάνουν ε, ε, τι γίνεται με τις ε, επενδύσεις, τι γίνεται με τις επενδύσεις. Άρα το πρώτο και βασικό θέμα είναι το αν υπάρχει διαφάνεια. Επίσης, με δεδομένο τον ανταγωνισμό στα χρηματοοικονομικά, θα πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία ολιγοπολίων. Να αποφύγουμε επίσης τις συγκεντρώσεις στην χρηματοοικονομική αγορά. Επίσης, θα πρέπει η φορητότητα για κάποια προϊόντα να διευκολυνθεί οι ασφαλίσει ζωής, οι ασφαλίσεις υγείας, οι συντάξεις. Θα πρέπει να αναπτύξουμε την ψηφική αγορά και την τεχνολογική καινοτομία όσον αφορά τις υπηρεσίες ε, για τις πληρωμές. Να μην υπάρχουν επίσης διακρίσεις ανάλογα με τον τόπο διαμονής. Αυτά είναι τα ζητήματα, οι βασικές αρχές επί των οποίων τελικά συνέκλυνε οι απόψεις μας. Κάτι άλλο θέλω να πω ότι υπάρχουν ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τοποθετηθεί. Τι γίνεται επομένω με κάποια ζητήματα συγχρηματοδότησης, τι γίνεται, θα υπάρξει κάποιο είδους συγκεκριμένη νομοθεσία για τα υπόλοιπα ε, χρηματοοικονομικά προϊόντα retail banking, λιανικής. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις προτάσεις αναμόρφωσης του τραπεζικού συστήματος σε σχέση με την συνθήκη υπαριθμών 3 της Βασιλείας. Βέβαια, επικεντρώσαμε στην προσοχή μας στο προκείμενο θέμα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και πέρα από το συγκεκριμένο. Πώς θα υπάρξει κάποιο είδου ασπίδα για το ε, σύστημα, γιατί είδαμε τι χτυπήματα δέχτηκε από το 9 και μετά. Μην χάσουμε το τρένο. Να μην ξαναβυθιστούμε σε μια άλλη χρηματοοικονομική κρίση, σε ένα άλλο τσουνάμι. Άρα θα πρέπει να το προσέξει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω τα πράγματα ορίμασαν για να δώσει κάποιες αντιθυντήρες γραμμές. και να προστατεύσει έτσι τους καταναλωτές, τους ε, αποταμιευτές οι οποίοι ακόμα διατρέχουν τρομερούς κινδύνους. Κάτι άλλο τώρα. Λέμε να έχουμε συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού και ε, κανόνες παιχνιδιού δίκαιους, αλλά έχουμε τόσες και τόσες ανισότητες. Άρα αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε και εδώ εμείς ίσως κατεβάσουμε κάποια τροπολογία υπομορφή επίκριση του κειμένου, γιατί εδώ έχουμε κάποιες ε, διαφορές μεταξύ των επιμέρους ε, χωρών. Άρα θέλουμε να καταλήξουμε με κάποια στεγανή ρύθμιση. Ε, ευχαριστούμε πολύ, ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω άλλες να ζητούν το λόγο. Α, όχι, όχι. Ο Ράιν Χέιζ ζητεί το λόγο. Πολύ σύντομα θέλω κι εγώ να σχολιάσω και να ευχαριστήσω βέβαια τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα επί της πράσινης αυτής βίβλου. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί δεν έχουμε ενιαία αγορά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό των λιανικών υπηρεσιών. Υπάρχουν διαφορές στη γλώσσα, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στη μία αγορά και την άλλη, διαφορετική διανομή, διαφορετική, διαφορετικός τρόπος με τον οποίο φτάνουν στην αγορά τα προϊόντα. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο εμεί δεν είμαστε καλοί εδώ στην Ευρώπη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το να ε, κοιτάμε και να διαλέγουμε ό,τι μας συμφέρει περισσότερο, ό,τι είναι καλύτερο για μας. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό. Η ενδιάμεση δεν έχουν τα κέρδη που θα μπορούσαν να έχουν και ο ανταγωνισμός είναι στοιχείο κλειδί εδώ. Αν δείτε τις υποθήκες στη χώρα μου. 2% παραπάνω από ό,τι σε άλλες χώρες ε, μέλη. Γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο φιλόδοξοι. Και το λέω επίτηδες έτσι το διατυπώνω, γιατί φυσικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για μια εναρμονισμένη προσέγγιση δεδομένων των διαφορών που υπάρχουν. Και το μόνο που έχω να πω πάντως στον εισηγητή και τους σκιώδες είναι ότι πρέπει να είμαστε όσο φιλόδοξοι μπορούμε να είμαστε. Να βοηθήσουμε τον κόσμο στον τομέα των λιανικών υπηρεσιών. Έχουμε τώρα μια αρχιτεκτονική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε συστημικό κίνδυνο. Το ίδιο και για την ε, Τραπεζική Ένωση, παρόλο που παραμένουν κάποια ζητήματα. Όμως αυτό που έχουμε κοιτάξει λιγότερο μέχρι τώρα είναι αυτό ακριβώ ο τομέα. Και αυτό είναι που νοιάζει πολύ τον κόσμο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά αυτή την πράσινη βίβλο, Πρόεδρε. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Άλλο κανεί. Τότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Παρακαλώ. Πέλε, όχι βέβαια όπως ο ποδοσφαιριστής, έτσι. Σχεδόν, σχεδόν, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως είπαν πολλοί εδώ, υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός το Δεκέμβριο με την πράσινη βίβλο. Και εμείς αντιμετωπίζουμε τώρα την πρόκληση να διατηρήσουμε αυτόν τον ενθουσιασμό. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, να προτείνουμε ένα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο δράσης. Το να βάσει κανείς στο κέντρο τον καταναλωτή σημαίνει συγχρόνως ότι πρέπει να κοιτάξει ποιες πραγματικά είναι οι ανάγκες του καταναλωτή και να φροντίσει ο κλάδος να ανταποκριθεί. Προς το παρόν αναλύουμε τις απαντήσεις που πήραμε στις προτάσεις της Πράσινης Βίβλου και από διάφορες ομοσπονδίες και από αρχές και από καταναλωτές πολλοί από εσά συμμετείχαν. Ο εισηγητή, κάποιοι σκιώδε εισηγητέ που συμμετείχαν και στη διάσκεψη που οργανώσαμε ενεργά. Σημειώσαμε ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να αποτελέσει μόχλευση για να έρθουν τα εμπόδια που έχουμε μέχρι τώρα στην εσωτερική αγορά και την οικονομική αγορά, που είναι περισσότερο στα χαρτιά παρά πραγματικότητα. Φυσικά θέλαμε το feedback από τους καταναλωτές και από όλους όσοι απάντησαν και όσον αφορά την οδηγία για τις πληρωμές όπου δεν υπήρχε το διασυνοριακό στοιχείο όσον αφορά την οδηγία υπηρεσιών πληρωμής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση, στα οποία θα εντρυφήσουμε περισσότερο. Την έκθεση του Κοινοβουλίου την βλέπουμε σαν συνεισφορά στη διαβούλευση αυτή υπάρχουν ακόμα περιθώρια να λάβουμε υπόψη μας αυτά που μας είπατε εδώ σήμερα, όπως για παράδειγμα το Green Finance, την πράσινη πτυχή του ζητήματος. Θα φροντίσουμε και για πρωτοβουλία όσον αφορά την ε, σήμανση. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ναι και όντω ελπίζω να διατηρήσετε ζωντανό τον ενθουσιασμό. Λοιπόν, όλε τι έχετε να συμπληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ για τις απόψεις σας σήμερα το απόγευμα. Και νομίζω ότως ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος. Δεν μπορεί να καθόμαστε και να περιμένουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Πιστεύω ότι τώρα πρέπει να δράσουμε. Αν δεν κάνουμε τίποτα για να φτιάξουμε αυτή την εσωτερική αγορά, θα μας προλάβουν άλλοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν νομοθεσία για να παρακολουθήσουμε το ζήτημα, να ενισχύσουμε τη θέση των καταναλωτών. Σημείωσα όσα είπαν οι σκιώδες, είναι σαφή. Θα τις κοιτάξουμε λοιπόν όλες αυτές τις ιδέες. Προσπαθώ να πετύχω συνένεση όπως σας είπα. Και από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπαν σήμερα οι Σκιώδης είναι ότι χρειαζόμαστε καλή δουλειά ώστε το ζήτημα αυτό να προβλεφθεί περισσότερο. Μα πόσο μπορούμε να περιμένουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε πολύ. Πρέπει να αρχίσουμε να περάσει η νομοθεσία ώστε να ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ε, ενιαία αγορά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση που θα μας οδηγήσει προς το μέλλον. Η αγορά καθημερινά αλλάζει, συνεχώς. Τίποτα δεν μένει ακίνητο. Οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε και πάλι το λόγο και προσβλέπω σε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Πραγματικά ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ χρήσιμη πρόταση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους όσοι συμμετείχαν στην ε, συζήτηση. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. 13 Ιουνίου περιμένουμε το σχέδιο έκθεσης. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 28 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Θα εξεταστούν οι τροπολογίες στις 31 Αυγούστου και θα ψηφίσει η Επιτροπή μας στις 29 Νοεμβρίου. και μάλλον στην πρώτη ολομέλεια του Νοεμβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία. Ελπίζω να σας κάνει αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ωραία, τελειώσαμε με αυτό το σημείο. Ωραία. Σημείο 5 στην ε, ημερήσια διάταξη, υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα. Πολύ σημαντικό. Έχουμε και άλλα ζητήματα που μοιάζει ο τίτλος αλλά είναι σε διαφορετικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Θα δώσω το λόγο αντί για τον Τάριους Ροζάτη στον ε, Λούδι Γουντεμάγερ. Σε ευχαριστώ πολύ Μάρκος να σας πω Ποιε είναι οι πληροφορίες που μου για το θέμα ο κ. Ροζάτη όπως γνωρίζετε για το θέμα αυτό εμείς έχουμε συμβουλευτικό ρόλο απόφαση θα λάβει το Συμβούλιο. Και όπως γνωρίζετε πριν από μήνες, δυστυχώς, το Συμβούλιο ήδη συνεφώνησε να ληφθεί η πολιτική απόφαση για το θέμα. Έτσι έχει η πραγματικότητα. Βεβαίως και θα υπάρξουν ε, συνέπειες. Πάντως ο κ. Ρωσάτη θέλει να τονίσει ότι η συνεργασία ήταν πάρα πολύ θετική και αποτελεσματική μεταξύ αυτού και των σχεδόν και επίσης έχουμε την ε, τελική ψήφιση του κειμένου τον Μάιο. Ελπίζει όπως η ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρόκειται να συνεχίσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενημερώνει ότι η σταλή επιστολή στο Συμβούλιο για την κατάσταση. Μέχρι σήμερα το Συμβούλιο δεν απήντησε. Αυτό βέβαια είναι απογοητευτικό. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό για την συνεργασία μας στο μέλλον όσον αφορά τα φορολογικά. Οπότε θα πρέπει, λέει ο κ. Ζωσάτη, να συμβαστούν το Κοινοβούλιο τα θεσμικά όργανα και να υπάρξει καλύτερη συνεργασία, ελπίζει, στο μέλλον. Τώρα επί της ουσίας. Από ό,τι γνωρίζουμε, πρόκειται για την πρώτη τέτοια οδηγία η οποία αφορά το πρόβλημα BEPS ΩΣΑ για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ε, βάσει του, των προτάσεων Μοσκοβής. Έχουμε 140 περίπου τροπολογίες και από τις οποίες προέκυψαν 10 συμβαστικές. Οι περισσότερες πολιτικές ομάδες συνεφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταπολεμήσει φόρο φοροδιαφυγή και φοροποφυγή με νέο μέτωπο και να υπάρξει επομένω ε, αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Οτροπή είναι ο φύλακα των συνθήκων, αλλά επίση θα πρέπει και να υποπτεύσει την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής. Άρα θα παρουσιάσει κάποιε προτάσεις σε Συμβουλίο και Επιτροπή και Συμβουλίο και Κοινοβούλιο όσον αφορά την οδηγία. Τώρα, έχουμε δύο ουσιαστικά ζητήματα τα οποία τα συζητήσαμε και σύμφωνα τον κυριο ρασατη Ρωσάτη πρώτα-πρώτα είχαμε τα 750 εκατομμύρια ως κατόφλι. Κάποιες πολιτικές ομάδες θέλουν μικρότερο κατόφλι. Αλλά ο εισηγητής θεωρεί ότι μια τέτοια αλλαγή θα δημιουργούσε άνισες συνθήκες για κάθε χώρα γιατί θα υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά τις χώρες που έχουν συμμετάσχει στον ΠΕΠΣ μέχρι τώρα. Σύμφωνα με του υπολογισμού του ΟΣΑ, αυτό το κατόφλι καλύπτει περίπου 90% των εταιρικών εσόδων. Επίσης, υπήρξε θέμα πεδίου εφαρμογής θεωρεί ο εισηγητής του πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το CPCR κάτι το οποίο προσφυλάστηκε πριν από δύο εβδομάδες από την Επιτροπή πάντως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του ΩΣΑ όσον αφορά ε, τους δίκαιους κανόνες παιχνιδιού και ανταγωνισμού. Θα πρέπει επομένω να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ διαφάνειας και παρανόμων πρακτικών. Να μην χτυπήσουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες, να έχουμε ένα περιβάλλον υγιές που να βοηθά τη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και τις επενδύσεις. Λούντεκλε πρόεδρε, ευχαριστούμε. Και τώρα, οι Αντί του κ. Μορέλ, έχει το λόγο ο κ. Μπαγιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συγχωρήστε τον κύριο Μορέλ. Ανταυτού, εγώ θα σας πω πώς βλέπει τα πράγματα. Θα σας διαβάσω το σημείωμα του. Ένα από τα καλά της δημοσιότητας ε, που είχαμε με τα Panama Papers ήταν ότι έχουμε αυτές τις αναφορές και διεκθέσεις ανά χώρα και επειδή πάρα πολλά χρόνια υπήρχε ένα πρόβλημα τώρα όμως είναι πάρα πολύ θετικό γιατί βλέπουμε ότι θέλουν τώρα να προχωρήσουν προς αυτό το μέτωπο και με διαφάνεια τα δεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη γιατί βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που είναι το να εφαρμοστεί η φορολογική νομοθεσία. Χρειάζεται όμως αυτό να γίνει με αποτέλεσμα θεμητών ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Έχουμε ένα άρθρο τη συνθήκη, που είναι η βάση των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά την εσωτερική αγορά. Επομένω, αύριο πριν την ψηφορία θέλει ο κ. Μορέλ να λάβετε υπόψη ότι δεν θέλουμε να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερο τζίρο, δηλαδή, δεν είναι σπρακτική η στόχη, αλλά θέλουμε να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερε πολιεθνικέ επιχειρήσει και έτσι να υπάρξουν ομοιόμορφε συνθήκε μεταξύ εθνικών εταιριών και πολυεθνικών στην ενιαία αγορά. Και θεωρεί επομένω ο, ο Μορέλ ότι δεν κατέληξαμε σε καμία συμβαστική συνεννόηση με τον εισηγητή και ο καθένας κράτησε την άποψή του. Έχουμε τώρα τέσσερι προτεραιότητε. Θεωρούμε ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να τις προτάξει αυτές τις ιδέες να μην είναι μόνο ε, συμβουλευτική γνώμη του. Άρα θα κάτι θα πρέπει να γίνει για τα φορολογικά. Οι προτεραιότητα μας είναι εξίσου. Όπως όλοι είπαμε ότι θα πρέπει να, να θεωρηθεί η οδηγία για τους μετόχους θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις σε όλες τις πολυεθνικές, σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και είπαμε θα πρέπει να καλύψουμε τις ε, θέσει που έχουν 250 εργαζομένους και 40 Εκατομμύριο τζίρο. Θα πρέπει επομένω να δούμε το πώς θα καταπολεμήσουμε το φορολογικό dumping και θα υπάρξει αρκετή πίεση στα κράτη-μέλη μόνο εάν εφαρμοστεί το CPCR για όλες τις πολυεθνικές που έχουν έδρα στην, ε, και λειτουργούν στην Ευρώπη. Και να υπάρξει επομένω αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών των κρατών μελών. Ακόμα ε, δεν έχουμε ευρωπαϊκό ορισμό για το τι θα πει μόνιμη εγκατάσταση πολυεθνική, άρα δεν θα πρέπει αυτό να είναι κριτήριο. Άρα, να δούμε τι θα γίνει την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων. Ανταλλαγή όλων των στοιχείων για να μην υπάρξει φοροαποφυγή. Επίσης, να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία, όπως τις κρατικές ε, ενισχύσεις ε, σε κάθε χώρα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ενημέρωση για αυτά τα στοιχεία γιατί έχουμε την οδηγία DAC. Και επίσης θα πρέπει να δούμε αν ε, ισχύουν οι εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις σε σχέση με την αποχρεωτική ανταλλαγή στοιχείων. Κάθε μέρα προχωρούμε στον αφορά τα και την Ερευνητική Επιτροπή από τη μία μεριά έχουμε την εθνική κυριαρχία, από την άλλη μεριά έχουμε και τη δημοκρατία. Άρα θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εάν δεν αλλάξει τίποτα στο κείμενο, δεν θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου. Θα τους απογοητεύσουμε. Είδατε τι έγινε και με το εμπορικό απόρριτο και την ψηφοφορία στην τελευταία ολομέλεια. Άρα και για το Panama Papers θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλες οι μεγάλες πολυεθνικές όχι μόνο το 10% θα πρέπει να καλυφθούν από αυτή την αρχή της ε, υποβολής έκθεσης ανά χώρα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Η κυρία Λέρνερ έχει τον, το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει και το γεγονό βεβαίω ότι αναζητούσε και αναζητεί συμβασμό και να ευχαριστήσω και τους ε, συναδέλφου για την συνεργασία. Νομίζω πω έχουμε επιτύχει μια χρυσή τομή η οποία αντικατοπτρίζει θα έλεγα τις απόψεις όλων των ομάδων στο Κοινοβούλιο για να καταπολεμήσουμε την επιθετική φόρο αποφυγή και φορολογικό σχεδιασμό και τα προβλήματα που έχουμε με τη φορολογική βάση. Αυτό δημιουργεί κίνητρα για εκθέσεις αναχώρα, για την ανταλλαγή πληροφοριών και χάρη στις ε, εκθέσεις αυτές οι εθνικές αρχές πιθανότατα θα έχουν καλύτερα εργαλεία στην διάθεσή τους έτσι ώστε οι πολυεθνικές να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υποχρεώσεις τους. Επίσης ε, και η πρόταση για τις αναφορές αναχώρα στηρίζεται στις ε, προτάσεις του ΩΣΑ. Γεγονό είναι πως ε, τα φαινόμενα αυτά είναι διεθνή και χρειάζονται διεθνείς λύσεις. Κατά την άποψή μου θεωρώ πως η πρόταση αυτή είναι ένα ημίμετρο όσον αφορά την ε, διαφάνεια και την αύξηση της διαφάνειας και τα κατόφλια τα οποία υπάρχουν επίσης το πεδίο εφαρμογής ε, και το χρονοδιάγραμμα. Θεωρώ πως θα έπρεπε να έχουμε θέσει στόχους πολύ πιο φιλόδοξους από αυτούς του ΩΣΑ. Όπως ξέρουν περισσότερες χώρες ε, του ΩΣΑ έχουν δεσμευτεί στις ε, σχετικές κατευθυντήρες γραμμές, αλλά βεβαίω λυπούμεθα για το ότι μια χώρα η οποία ήταν τελευταία πολύ στις ειδήσει δεν έχει δεσμευτεί. Αλλά όπως είπα στην αρχή είμαι αρκετά ικανοποιημένη με τη δουλειά του κυρίου Ροζάτη και ελπίζω να συνεχιστεί η επικοδομητική συνεργασία. Είναι προς το συμφέρον όλων μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο φιλελεύθερους, την κυρία Φανίεν Γόιζεν ε, και βεβαίως την συγχαίρουμε για την νίκη στο Ρότερνταμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα τα, θα τα διαβιβάσω. Ε, ναι βεβαίως, αλλά πρέπει να προκριθείτε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ροζάτη για τα καλά του λόγια, όχι μόνο για την καλή δουλειά που έκανε, όχι μόνο για τις διαπραγματεύσεις αλλά και για τις συμβαστικές προτάσεις οι οποίες είναι θετικές και μπορούμε να τις ε, στηρίξουμε. Καλό είναι το ότι όλοι είμαστε υπέρ του να γίνει υποχρεωτική η ανταλλαγή πληροφοριών και αυτόματη και να βασίζεται σε ενιαίους ορισμούς και βεβαίως αμοιβαιότητα. Ο κύριος ε, Ροζάτη στην ε, έκθεσή του έχει πει πως θα πρέπει να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα αυτών των αυτομάτων ανταλλαγών ε, και συμφωνούμε πλήρως και προσπαθήσαμε να το ενισχύσουμε. Έχουμε βάλει κάποιες τροπολογίες και ζητάμε όχι μόνο να μας λένε ποιες ήταν, πόσες ήταν οι ανταλλαγές, όχι μόνο τον αριθμό τους, αλλά και ποιοτικά στοιχεία, ποιο ήταν το αποτέλεσμα και τι γίνεται τελικά. Και χαίρομαι τώρα που σε μια συμβιβαστική πρόταση λέγεται ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο και για τον αριθμό και για το αποτέλεσμα. Γιατί δεν θέλουμε να είναι κάτι το οποίο θα μείνει στα χαρτιά και δεν θα το ξανακούσουμε ποτέ. Ένα τελευταίο αίτημα λοιπόν προς τους συναδέλφους μας. Μία άλλη τροπολογία που έχω συντάξει δεν έχει γίνει δεκτή και αφορά την αναθεώρηση. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή κάποια αναθεώρηση του κανονισμού. και έχω υποβάλει μια τροπολογία που λέει πως μετά από τρία χρόνια θα πρέπει να ξαναδούμε αν εφαρμόζεται σωστά, εάν μας δίνει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, οπότε θα ήθελα να ξαναδείτε να, να ξαναδούμε και να αξιολογήσουμε τον κανονισμό αυτό σε τρία χρόνια. Αυτά κύριε Πρόεδρε για την ώρα. Σας ευχαριστώ κόρα. Δεν βλέπω κάποιον από την ΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, είμαι εδώ για εξ ονόματος του σκιώδος ε, εισηγητού ο ε, σε σε πολλά με τον συγητή έχει και κάποιες τροπολογίες, εξπακούεται πως ε, είναι υπέρ της ε, μέγιστης δυνατής διαφάνειας για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις τις οποίες έχουμε δει. επίση στηρίζει τις εκθέσεις αναχώρα. Όμως έχει πολλές ανησυχίες με την πρόταση που λέει πως η Κομισιόν θα πρέπει να έχει ευθύνη και αν είναι με, υποχρεωτική, ή με υποχρεωτικό χαρακτήρα, έστω, αλλά δεν θα πρέπει να έχει τον τελικό λόγο και ευθύνη κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στους πράσινους. Δίνω λόγο στην κυρία Κέιτο. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρό η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, δεν είναι όμως ε, αυτό το οποίο θα θέλαμε οι εκθέσεις αναχώρα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, αλλά σε κάποια σημεία δεν θεωρώ πώ ε, είναι σωστή η θέση του Κοινοβουλίου. Το βασικό θέμα είναι το κατόφλι για το μέγεθος των εταιριών. Και εδώ πέρα και στην πρόταση της ε, Κομισιόν για τις εκθέσεις αναχώρα που βγήκε πριν από λίγες εβδομάδες έχουμε πολύ υψηλό κατόφλι για έναν τζίρο 750 εκατομμυρίων ευρώ. Ως πράσινοι θέλουμε το κατόφλι να ευθυγραμμιστεί με το κατόφλι των μεγάλων επιχειρήσεων όπως ορίζονται στην οδηγία περί λογιστικών, όπου ο τζίρος είναι τα 40 εκατομμύρια. Δεν ήμασταν οι μόνοι που είχαμε αυτή την θέση. Είχαμε στήριξη και από την Κόσο Σελδημοκράτες η FTD και του φιλελεύθερου όμω, ε, αποφάσισε ο εισηγητή να μην το βάλει στην έκθεσή του. Αυτό με απογοητεύει, οπότε θα ήθελα να ζητήσω από όλε τι πολιτικές ομάδες να τονίσουν αυτέ τι τροπολογίε τους ε, καταλόγους και να υπερψηφίσουν τι τροπολογίε 133 έω 166. Επίση, το είπαν ήδη το Κοινοβούλιο απλά γνωμοδοτεί καθώς το Συμβούλιο έχει φτάσει σε μια άτυπη συμφωνία με την Κομισιόν. Όμως θεωρούμε πως υπάρχει ανάγκη να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι ως εκπρόσωποι των λαών της Ευρώπης ε, θέλουμε ένα πιο ισχυρό πλαίσιο από αυτό το οποίο καθορίζει ο ΣΑΝ είναι να παίρνουμε στα σοβαρά την διαφάνεια. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πιο σοβαρή θέση για να μην αποφύγουμε ακριβώς ε, την ε, εντύπωση η οποία υπήρχε με το προηγούμενο που δημιουργήθηκε με τη Συμφωνία Κομισιών και Συμβουλίου που παρέκαμψε τα Ε, δημοκρατικά όργανα. Επίσης υπάρχουν τροπολογίες 45 και 128 που αφορούν την αρχή της αμοιβαιότητα ε, και την φορολογία στην πηγή με τις χώρες ε, στις οποίες δεν ανταλλάσσουν αυτομάτως στοιχεία. Ως πράσινοι το έχουμε ζητήσει αυτό μετά τις αποκαλύψεις στα έγγραφα του Παναμά και άλλες περιπτώσεις όπου πηγαίνουν τα μετρητά σε υπεράκτιους λογαριασμούς και έτσι Νομίζω πως ε, μπορεί εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο φιλόδοξη από τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης με απογοήτευσαν οι φόβοι που εξέφρασαν διάφοροι συναδελφοί για ζητήματα εμπιστευτικότητας εμπορικών μυστικών. Δεν θα πρέπει αυτό να μπλοκάρει την ε, πρόοδο. Οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν στα δεδομένα αναχώρα δεν περιέχει εμπορικά μυστικά. Και δεν θα πρέπει άρα να το χρησιμοποιούν ως δικαιολογία οι εταιρείε το Συμβούλιο διέγραψε την αναφορά στο άρθρο 17.4, ενώ η τροπολογία μας η 75 το τονίζει αυτό. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες για δευτερογενείς αναφορές, ε, για κάποια επικουρικότητα και βεβαίως τις ανταλλαγές στοιχείων με αναπτυσσόμενες χώρες και κυρώσεις για την μη υποβολή αναφορών, αν είναι να έχει κάποια ουσία αυτό το πράγμα. Οπότε θα θέλαμε να ζητήσουμε από τους συναδέλφους να εξετάσουν αυτές τις τροπολογίες που θεωρούμε ότι ενδυναμώνουν την πρόταση. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Μπίμπλ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα φορολογικό σύστημα που πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό του οι επιχειρήσει. Αυτό ήταν ε, προτεραιότητα ανέκαθεν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ενίσχυση τη διαφάνεια λοιπόν αφενό ανάμεσα στι φορολογικέ αρχέ ε, αφετέρου προ το ευρύτερο κοινό είναι ζωτική σημασία για να δημιουργηθεί ένα πραγματικά δίκαιο σύστημα. Και ένα από τα μέτρα που δημιουργήθηκαν ήδη από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς ήταν αυτή η αυτόματη ανταλλαγή πληροφορών όσον αφορά του φορολογικού διακανονισμού. Ευχαριστώ λοιπόν την Επιτροπή σα και γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καλή συνεργασία που είχαμε, παρόλο που το χρονοδιάγραμμα ήταν πάρα πολύ σφιχτό. Και ήταν έτσι σφιχτό, διότι όλοι πιστεύουν ότι πρέπει γρήγορα να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα, να μην χάνουμε χρόνο Και η συγκεκριμένη πρόταση προσφέρει στις φορολογικές αρχές τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να μπορέσουν να αναλύσουν οι ίδιες καλύτερα την κατάσταση. Οι πληροφορίες αυτές, επί του παρόντος, δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις φορολογικές αρχές. Βοηθάει τις φορολογικές αρχές να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και να προβούν σε ελέγχους, φορολογικού ελέγχους. Άρα θα υπάρξει σίγουρα βελτίωση για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Δεν είναι στόχος της πρότασης αυτής να προσφέρει στο γενικό, στο γενικό κοινό περισσότερες πληροφορίες για να ελέγχει. Όχι, υπάρχει μια διαφορετική πρωτοβουλία που θα καλύψει αυτό το ζήτημα. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση αυτή ήταν να μεταφέρει τη δράση που συμφωνήθηκε σε επίπεδο ΩΣΑ κομμάτι-κομμάτι. Και είναι σημαντικό αυτό για μας, διότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν δημιουργούμε διαφορετικά επίπεδα κοινοποίηση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνοχή στην αντιμετώπιση οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται πρέπει να είναι επίσης συγκρίσιμες. Κύριος στόχος μας λοιπόν στην άσκηση αυτή ήταν να δημιουργήσουμε ίσους όρους ανάμεσα στις ε, ευρωπαϊκές ε, πολυεθνικές και τις μη ευρωπαϊκές πολυεθνικές. Και έχει αγωνιστεί σκληρά προς αυτό το σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πετύχαμε ότι με τον δευτερεύοντα αυτό μηχανισμό, όπως αναφέρθηκε, όλοι οι πολυεθνικοί όμιλοι που δεν είναι ευρωπαϊκοί αλλά που δραστηριοποιούνται μέσα στην Ευρώπη υποβάλλονται στο CBCR, άρα ενημερώνονται φορολογικές αρχές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι μια καλά ισορροπημένη πρόταση. Για τα όρια. Όσον αφορά τα όρια που εκφράσατε την ανησυχία, ακολουθούν τα συμφωνημένα σε επίπεδο ΟΟΣΑ και όσον αφορά το ΠΕΠΣΤΗ Η διάβρωση βάση και μεταφορά κερδών. Τα 750 εκατομμύρια που αναφέρονται ως ποσό έχει να κάνει με ομίλους και μέσα σε έναν όμιλο μπορεί να υπάρχουν διάφορες οντότητες θυγατρικές με χαμηλότερα όρια από 750 εκατομμύρια. Είναι το συνολικό ποσό που μετράει. Δεν ήταν σκοπός μας να καλύψουμε ένα ποσοστό του τζίρου, αλλά να δείξουμε ότι το όριο, παρόλο που φαίνεται υψηλό, καλύπτει πάνω από το 90% του συνολικού εισοδήματος. Αν χαμηλώσει αυτό, τότε για μερικές περιπτώσεις δεν θα καλύπτουμε μεγαλύτερο επίπεδο σε ποσοστό εισοδήματος. Γι' αυτό και εδώ πιστεύουμε ότι πολύ καλά ακολουθεί την αναλογικότητα η πρόταση αυτή. Για το απόρριτο, ναι, διαγράφει το 74, αλλά η αιτιολογική σκέψη λέει ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται υπό την πρόταση αυτή δεν είναι απόρριτες. Όπως είπα, το δημόσιο στοιχείο αντιμετωπίζεται με διάφορες προτάσεις που θα συζητηθούν στο εγγύς μέλλον. Πιστεύουμε ότι η έγκριση της πρότασης αυτής λοιπόν με τη βοήθεια της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βοηθήσει τις φορολογικές αρχές να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται. Επίσης θα υπάρχει και ένα ισορροπημένο βάρος κατά κάποιο τρόπο για όλες ε, τις πολυεθνικές και αυτές που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές που είναι εκτός. Θα υπάρχουν ίδιες απαιτήσει. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος, προκειμένου να πετύχουμε τη διαφάνεια, το γνωρίζετε όλοι. Πρόκειται για ένα βήμα μόνο που έχουμε κάνει. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα προσβλέπω σε συνέχιση της επικοδομητικής συνεργασίας που έχουμε μεταξύ μας. Και σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Λιούτεκ, εσύ που αντικαθιστά τον εισηγητή, θες να προσθέσεις κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές. Ελπίζω και εγώ η συνεργασία αυτή στην οποία αναφέρεται ο εκπρόσωπο τη Επιτροπής να επιτευχθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι ήταν ακριβώ έτσι. Καλώς, λέει Ευχαριστώ πολύ και τον συγκητή και όλους σας. Τώρα, όπω έχει συμβεί και με άλλε νομοθετικές προτάσεις, το Συμβούλιο καταφέρει να φτάσει σε μια πολιτική συμφωνία και περιμένει εμά. Όπως είπε όμως και ο κύριος Μπίπ, δεν είμαστε στο τέλος της διαδικασίας. Οπότε ας φροντίσουμε να περάσουμε περισσότερο τα πράγματα. Προβλέπετε η ψηφοφορία αύριο. Αύριο ψηφίζουμε από τις 11 και 45 μέχρι τις 12 και 30. Να έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και εγώ ξεχάσω, λέει ο πρόεδρος. Στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε στην πρώτη σύνοδο του Μαΐου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για το σημείο 7. Θα δώσω το λόγο στον αντιπρόεδρό μας για την Προεδρία. Okay, dear colleagues, um, before we start... Συνάδελφοι, πριν συνεχίσουμε, πρέπει να σας πω ότι μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε τη συνεδρίαση για περίπου μισή ώρα κάποια στιγμή αργότερα. Αργότερα, μετά από αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα. Και θα ξαναρχίσουμε στις 6. Άρα στις 6 θα συζητήσουμε το επόμενο θέμα που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα για 20 λεπτά μισή ώρα θα πρέπει να διακόψουμε μεταξύ του τωρινού θέματος και του θέματος των ΜΜΕ. Και τώρα πάμε στο θέμα υπαριθμών 6. Πρόσβαση στην χρηματοδότηση των ΜΜΕ και αύξηση πολυμορφίας της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγόρων. Σήμερα έχουμε τις 249 τροπολίες που θα εξετάσουμε. Οπότε πρώτα πρώτα θα μας μιλήσει ο εισηγητής Ότμαρ Κάρας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις τροπολογίες. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να τονίσω πως ε, θέλουμε ευρία στήριξη όλων των βουλευτών για αυτή την έκθεση γιατί θεωρούμε πως ε, πρέπει να υπάρχει μια σαφής ε, θέση για το θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί έτσι θα χρηματοδοτηθεί η πραγματική οικονομία και θα ενισχύσουμε την ε, Κεφαλαιακή Ένωση. Βλέπετε λοιπόν δεν θα χωρίσω τις ε, τροπολογίες, ε, δεν τις έχω χωρίσει ε, κομματικά αλλά θεματικά στις συμβαστικές τροπολογίες. Ε, νομίζω πως τις καλύτερες ιδέες θα τις κάνω δεκτές. Μίλησα και με τους χειώδεις ηγητές πριν λήξει κάνει προθεσμία για τις ε, τροπολογίες για να καταλήξουμε σε τροπολογίες οι οποίες θα εμβαθύνουν και θα συμπληρώσουν την έκθεση και να μην γίνει η έκθεση μια έκθεση στην οποία θα γράφει ο καθένας ό,τι θέλει και πράγματα τα οποία καλύτερο, καλύτερα καλύπτονται αλλού. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει βάση για μια συζήτηση και λόγω του αριθμού των τροπολογιών βλέπουμε πως ε, από τον διαχωρισμό με βάση το μέγεθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι και τις ε, περιφερειακές ιδιαιτερότητες υπάρχει ανάγκη για μεγάλη συζήτηση. Θα προτείνω λοιπόν ανάλογα και θεματικές συμβιβαστικές ε, τροπολογίες για ένα καλύτερο ορισμό και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά την χρηματοδότησή τους τώρα θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και τις τροπολογίες των ε, συναδέλφων για να πω πως ε, θα πρέπει να είναι διασφαλισμένη χρηματοδότηση σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων. Πέρα από τις κλασικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όμως δεν θα πρέπει να ξεκινάμε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις και ειδικά εδώ πέρα οι περιφερειακές τράπεζες παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια στις μικρομισές επιχειρήσεις από ό,τι κάνουν μέχρι στιγμής. Όμως είναι σαφές πως χρειάζεται και μια διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης. Μέχρι και περισσότερο επιχειρηματικό κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε καμία πηγή. Επίσης ε, είναι σημαντικό το να υπάρχει ο λεγόμενος βαθμός διευκόλυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έγινε πρόσφατα και μια συζήτηση στην Ολομέλεια. Επιπλέον είχαμε συμφωνία με τους χειοδησηγητές πως θα πρέπει να στηρίξουμε καλύτερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις ε, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα πρέπει να παρεμποδίζονται και εθνικές ε, πρωτοβουλίες. Χαίρομαι πως υπάρχουν πολλές τροπολογίες για μείωση της γραφειοκρατίας, για δικαιότερη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για καλύτερο ορισμό της αναλογικότητας, ε, τις οποίες θα ομαδοποιήσουμε. Σημαντικό είναι λοιπόν η συζήτηση αυτή να γίνει χωρίς ιδεολογικές παροπίδες όμως. Θα ήθελα να πω πως ε, οι συζητήσεις για τον τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης ή της ε, διαμόρφωσης ε, της τιτλοποίησης STS είναι κάτι το οποίο θα απορρίψω εδώ πέρα γιατί ε, υπάρχουν ξεχωριστές νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες εδώ πέρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οπότε δεν χρειάζεται να γίνει παράλληλη συζήτηση στο θέμα αυτό εδώ. Τα θέματα αυτά πηγαίνουν ε, στα αντίστοιχα νομοθετήματα τα οποία είναι επιτάπητος και όχι σε αυτή την έκθεση. Επίσης αυτονόητο Υπήρχαν κάποια πράγματα που έπρεπε να συζητήσουμε, υπήρξαν κάποιες φωνές για έναν ενιαίο αριθμό μητρώου μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή επιθυμία η Κομισιόν να βοηθήσει με κάποια προγράμματα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να κάνουν το άλμα σε άλλες υπήρους. Είμαι σίγουρος πως ε, θα μπορέσουμε να έχουμε μια ισορροπημένη έκθεση τελικά. Πολλές τροπολογίες με βρίσκουν ε, σύμφωνο. Είναι πολλές όπως ε, σας είπα στον αριθμό. Δεν υπάρχουν μεγάλες αντιφάσεις μεταξύ τους. Τα θέματα στα οποία αφορούν είναι αρκετά περιορισμένα και βεβαίως όπως είπα θα διαμορφώσω κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους κοιόδησίτες και θα ήθελα να ζητήσω μια ανοιχτή έντονη συζήτηση και συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Υπάρχει τώρα ένα αίτημα της Άλντε να ακούσουμε τον κύριο Τόρε ο οποίο αντικαθιστά τον κύριο Ντεμπάκερ, γιατί θα πρέπει να φύγει. Δεν νομίζω να υπάρχει καμία αντίρρηση. Κύριε Τόιρερ, για την Άλντε. Ναι, σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, που μου επιτρέπετε να μιλήσω πρώτο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Κάρας, για την ε, έκθεση του. Το ανέφερε η έκθεση της... Ε, η συζήτηση της Ολομέλειας ε, νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι κάτι μας, ε, το οποίο μας οδήγησε σε αυτή την έκθεση για τη χρηματοδότηση και ακριβώς λέμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ο Φίλιπ Τεμπάκερ τώρα θα ήθελε να πει πώς επικεντρωνόμαστε ως ομάδα στην χρηματοδότηση από πολλαπλές πηγές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρούμε επίσης πως η συνταγή, μία συνταγή για όλους δεν μπορεί να ισχύσει. Υπάρχουν πολλές πηγές όπως είπαμε. Είπαμε πως ε, δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο ρόλος των τραπεζών 99% των επιχειρήσεων στην Ένωση είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, γύρω στα 25 ε, εκατομμύρια και βεβαίως να το συγκρίνουμε με τις χρηματαγορές που είναι η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης της ε, ΕΠΑ είναι κάτι το μη ρεαλιστικό. Παρόλα αυτά και εδώ πέρα βεβαίως είναι το δεύτερο σημείο το οποίο τονίζουμε πρέπει να ενισχυθεί ακριβώς ο ρόλος των χρηματαγορών στην χρηματοδότηση των μικρομισών επιχειρήσεων και εδώ πέρα παίζει μεγάλο ρόλο η καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε υποβάλει και κάποιες σχετικές τροπολογίες. Θεωρούμε πως η Ένωση των Χρηματαγορών χρειάζεται ένα σε νομικό πλαίσιο με κάποια σύγκληση. Δεύτερον, θεωρούμε πως και το θέμα των ε, κοιματαγορών. για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να μας απασχολήσει αυτή την έκθεση και τρίτον θα θέλαμε η Κομισιόν να υποβάλει μια ετήσια έκθεση που πρακτικά θα μας λέει ποια είναι η εφαρμογή των σχετικών ε, πρωτοβουλειών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Τόιρερ. Τώρα περνάμε στην κανονική σειρά των ομιλητών για τους σοσιαλδημοκράτες για τον Σαν Σιμών, ο Ιουκ Μπαγιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον αδερφό που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ τον κύριο Κάρας για το ξέρετο έργο του, για την έκθεση αυτή, αλλά και όλους τους συναδέλφους σοσιαλιστές. Όπως έχουμε ήδη πει, είμαστε ικανοποιημένοι δεν διαφωνούμε πλήρω με κανένα σημείο για τι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την άδεια της τραπεζικής Ευρωπαϊκή αρχής. Δεν ξέρουμε κατά πόσο το supporting factor μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων. Οπότε ρωτάμε κατά πόσο η Επιτροπή έχει υπολογίσει, έχει εκτιμήσει τον αντίκτυπο ε, στην περίπτωση που αυτό γίνει μόνιμο. Όπως λέει και ο κύριος Καρά στην ε, έκθεσή του, καταλαβαίνουμε τη σημασία των τραπεζών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως αυτές που είναι πιο απομονωμένες. Γι' αυτό και θέλουμε να προωθήσουμε το ρόλο των τοπικών τραπεζών. Να υπάρχει διαφοροποίηση, αν μη τι άλλο, ώστε να μπορούν να ευνεθούν ε, τα δάνεια. Η κατάσταση είναι διαφορετική και η κοινωνικο-οικονομική και η γεωγραφική, άρα και η αντιμετώπιση πρέπει να είναι διαφορετική. Να σκεφτούμε λοιπόν διάφορες, διάφορους τρόπους χρηματοδότησης, είτε με κεφάλαια επενδύσεων, είτε crowdfunding κλπ. Πρέπει να ισχύσει αυτό στην αγορά των κεφαλαίων και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ρυθμιστικές λύσεις για να διασφαλιστεί επίσης και η διαφάνεια και η σταθερότητα στη διδλοποίηση αλλά και η πρόσβαση στις μικρές τράπεζες. Όσον αφορά τώρα τις δημόσιες επενδύσεις, θέλουμε ενισχυμένες επενδύσεις από το δημόσιο τομέα και κυβερνητικά δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα θέλαμε η Επιτροπή να σκεφτεί και σχέδια όπως το Funding for Landing που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να δανείσουν στις τράπεζες, εφόσον αυτές δανείζουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μόνο τότε. Και να συγκεντρώσουμε πληροφορίες προς όφελος των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των διακρίσεων που γίνονται στην πρόσβαση, στη χρηματοδότηση. Και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι αυτό το θέμα έχει ενδιαφέρον και θεωρούν σημαντικό και οι συνάδελφοι. Ένα πρόγραμμα ε, χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λοιπόν είναι αυτό που χρειάζεται και να δουλέψουμε και για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός ε, τραπεζικού σχήματος για την ενημέρωση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν έχουν πληροφορίες για την χρηματοδότησή τους αυτή και να βελτιωθεί και το σύστημα εξωτερικής αξιοπιστίας και φερικιότητας. Θέλουμε λοιπόν να δούμε πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ούγκο, Ούγκο, για το ECR. Και εδώ πέρα κάποιος αντικαθιστά τον κύριο Όσοκ και κυρία Σούνμπερν. Ευχαριστώ δεν να τον συμπαθήσετε τον συνάδελφο, αλλά θα σα πω εγώ τι παρατηρήσει του για το θέμα που συζητούμε τώρα. Πρώτα πρώτα ευχαριστεί τον εισηγητή και ε, τονίζει ότι ο κ. Κάρας ε, Στέταξε πάρα πολύ αξιόλογο κείμενο. Οι περισσότεροι σκιώδε, Όπω θα μα συνάντησή του, είπα είναι υπέρ. Και ο Ζωζέ επίση είπε ότι ε, υπήρχαν και κάποιε προστριβέ Οπότε δεν θα πρέπει να σας εκπλήξουν. Όλες αυτές οι τροπολογίες που πρόκειται να υποβληθούν για την εκθέση πρωτοβουλίας εξηγεί ότι θέλουμε να έχουμε μια κοινή τοποθέτηση για τις ΜΜΕ πλευράς της ΕΚΟΝ. Όμως διαπιστώνεται ότι έχουμε ένα σωρό τροπολογίες που αφορούν την μακροοικονομική προβληματική, αλλά έχουμε και, άλλα ζητήματα, τα οποία είναι αντικείμενο άλλων εκθέσεων μας Τέλος πάντων, Έχουμε κατεβάσει κάποιε λίγε τροπολογίε και λέμε ότι δεν χρειάζεται υπερβολική ρύθμιση, πολυνομία, ε, χρειάζονται απλοί κανόνε. Αλλιώ θα χτυπηθούν οι ΜΜΕ και η ανάπτυξη και γι' αυτό το λόγο συμφωνεί όλε τι τροπολογίε που αφορούν αυτό ακριβώ το πρόβλημα όπω την 67 ε, και την 87. Επίσης ε, έχει κάποιες επιφυλάξεις για τις τροπολογίες που θέλουν πλήρη εναρμόνιση όπως ας πούμε Φερρυπίν την υπερθυμόν 35 θα έπρεπε επίση να υπάρχει ουδετερότητα όσον αφορά τα δύο φύλλα και θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα τα μακροοικονομικά, τα θέματα τη λιτότητα, την χρηματοδοτική κρίση, την τροπεζική ένωση κλπ. Θεωρεί ο συναδελφό ότι θα πρέπει σε αυτή την ε, ένωση να είμαστε όσο είναι πιο συγκεκριμένοι. Θα πρέπει να σεβαστούμε στι ΜΜΕ. Άρα δεν συμφωνεί με τι τροπολογίε που είναι εκτό θέματο αυτή τη οδηγία να πετύχουμε προ μια κοινή θέση από πλευράς ΜΜΕ στην ε, Ένωση των Κεφαλαιογορών και να υπάρξουν επομένω εναλλακτικέ για χρηματοδότηση των εταιριών στην Ένωση και άρα μην αρχίσουμε να μιλάμε για ε, ρυθμιστικά ζητήματα Ή για το Ίντις Και επίσης, όπως είπε ο συγητής, όταν άρχισε αυτή η διαδρομή, ο συνάδελφος θέλει αυτή η έκθεση να είναι συγκεκριμένη για αυτό το θέμα και για το συγκεκριμένο σκοπό. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ για την Γκουα, για την Γκουα δεν είναι εδώ. Α, την αντικαθιστά κάποιος, κάποια. Όχι. Δίνω απευθείας το λόγο στους πράσινους η συνάδελφος κάτω αντικαθιστά τον κύριο Λαμπέρ. Ε, ευχαριστώ. Να, και στα γερμανικά που τώρα, μάλλον το κατάλαβα. Ο Φιλίπ δεν μπορούσε δυστυχώ να έρθει να μα τα πει. Οπότε θα σα πω εγώ για την εφαρμογή τη συνθήκη τη Βασιλεία 3 συμφωνούμε με τον κύριο Κάρα και θεωρούμε ότι παρά το ότι ο Φιλίπ Λαμπέρ ε, θεωρεί ότι η οδηγία 4 ε, δεν θα ήταν ο καλύτερο τρόπο να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες τι ε, δραστηριότητε από τι ΜΜΕ γιατί είπαμε ότι το θέμα είναι η οδηγία αυτή για την κεφαλογική απέτηση να συνάδει με την Βασιλεία 3. Οπότε έχουμε την έκθεση του EBA. Οπότε είπαμε ότι δεν ωφελεί για καλύτερο δανεισμό προ τι ΜΜΕ γιατί ε, οι σχετικέ τραπεζε χρησιμοποιούν κάποια εσωτερικά μοντέλα για να καλύψουν τι κεφαλικέ του απαιτήσει και σύμφωνα με την EBA ε, είπαμε ότι τελικά δεν βγαίνει τίποτα ιδιαίτερο, δεν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και όπω λέει η έκθεση, θα πρέπει οι τράπεζε να εξυπηρετήσουν περισσότερο τι ΜΜΕ, να έχουν ε, κεφαλαιοποίηση τέτοια, ούτω ώστε να μην ε, χρεώνουν οι, ιδιαίτερα μεγάλες ε, προμήθειες. Θα πρέπει με τη χρηματοδότηση να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία και να μην γίνεται τροχοπέδι αυτή η ρύθμιση για την πραγματική οικονομία. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ανθεκτικότητα όταν υπάρχει κάποια κρίση και να βοηθούν ε, οι τράπεζες ε, την ώρα της κρίσης, να μην δημιουργούν μια κρίση. Οπότε το πρόβλημα αυτό είναι επίγον, θα πρέπει να άρουν οποιουσδήποτε φραγμούς για την προσβασιμότητα στον δανεισμό και να έχουμε τέτοια μοντέλα δανεισμού που να είναι φιλικά στις ΜΜΕ και αξίζει να δούμε ότι όχι μόνο οι μεγάλες ε, τράπεζες αλλά και οι μεγάλες εταιρείες ε, όταν τα πράγματα ζορίσουν ε, ε, στριμώχουν τις ΜΜΕ για τις προμήθειες, για, για την αποπληρωμή του δανείου οπότε τελικά δεν πιάνουν τόπο οι, οι νομοθεσίες για την σωστή οικονομική διακυβέρνηση, ή διαχείριση. Θα πρέπει να υπάρχουν καινοτόμες λύσεις φιλικές προς τις ΜΜΕ τον καιρό της κρίσης. Αυτό μπορεί για, για τους δανειστές, τους δανειζόμενους να υπάρχει κάποιο είδους εκμίσθωση εξοπλισμού αντί για την αγορά του αλλά για αυτό το είδος το, το leasing θα πρέπει να μπορέσουμε να άρουμε τους φραγμούς. Δεν υπάρχει μαϊκή συνταγή για την επιτυχία του στήματος και των ΜΜΕ. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η ρύθμιση δεν θα τις ωφελήσει τις ΜΜΕ, θα ωφελήσει κάποιες τράπεζες, θα ωφελήσει κάποιους ενδιάμεσους και όχι τον πολίτη. Επίσης, ρίξαμε ιδιαίτερο βάρος στο πώς θα υπάρχει ε, ένα σύστημα το οποίο να μην είναι, έχει γιγαντισμό αλλά ανταποκρίνεται στις πραγματικές ε, ανάγκες σύμφωνα με τους κανόνες διακυβέρνησης της Ευρωζώνης και ε, έτσι να έχουμε την σταθερότητα για την οποία, την οποία χρειάζονται οι ΜΜΕ με κρατικές επενδύσεις και κρατικά ομόλογα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει για δυνάμει του ορίζοντου και για το κόσμο να δει αν υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση των ΜΜΕ και επίσης να μπορέσει να στηρίξει τις ΜΜΕ από τη, τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής κρίσης. Κλείνοντας, να σας πω ότι ε, η χρηματοδότηση και ο δανεισμός από τις τράπεζες δεν θα πρέπει να είναι οι μόνες πηγές χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικέ λύσεις θα πρέπει να δοθούν κίνητρα προς τούτο και εμείς στις τροπολογίες μας με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορέσουν να καταλευθούν την ε, πύρα ε, του συστήματος της Ελβετίας του 34 που ακόμα ισχύει και στο οποίο έχουμε αναφερθεί. Εκεί έχουμε μια τράπεζα συμπληρωματικού ε, παράλληλου ε, συστήματος που βοηθά την κάθε δραστηριότητα των ΜΜΕ και είναι δυνατόν η επιχείρηση μπορεί να αγοράσει απευθείας η μία από την άλλη χωρίς να χρησιμοποιήσει τα... το ελβετικό φράγκο του πάντων και αυτό ωφελεί το ΑΕΠ. Ευχαριστώ. Για το... Η ευθυντή ο Μάρκο Τσάν αν είναι, εδώ. Δεν είναι και δεν υπάρχει κανείς άλλος από την κοινοβουλευτική ομάδα. Για το ΕΝΕΦ e επίσης κανείς. Οπότε περνάμε κατευθείαν στο KTI. Στέρντε Λάγκε λοιπόν, έχει ζητήσει το λόγο. Ωραία, θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να στήριξω την προσέγγιση του εισηγητή. Κάτι το οποίο βρίσκω ενδιαφέρον είναι ότι πάντα μιλάμε για τις απορριφθήσεις αιτήσει για πίστοση και κοιτάμε τις χώρες του κέντρου και της περιφέρειας και λέμε πως οι αιτήσει για δάνεια, οι οποίες έχουν μειωθεί περισσότερες χώρες περιφέρειας. Δεν είναι τόσο άσπρα μαύρα τα πράγματα όμως. Αν δούμε τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πράγματι έχουμε 40% των ε, αιτήσεων που απορρίπτονται, στις κεντρικές χώρες μόνο 15%, αλλά αν δούμε τη χώρα μου την Ολλανδία, το ποσοστό απόρριψης είναι 45%. Ψηλότερο από της Ιρλανδίας και της Ισπανίας. Χαμηλότερο από την Ελλάδα μόνο. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να γνωρίζω είναι ποιοι είναι οι λόγοι γι' αυτό. Στην ε, έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν έχουν απάντηση. Αν δούμε τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας Ολλανδίας επίσης δεν έχουν κάποια απάντηση. Οπότε θα ήθελα να δω ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί. Γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν είναι μόνο ένας ο λόγος. Βασικός οπωσδήποτε λόγος είναι η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανάπτυξη της Ένωσης, αλλά ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από αυτά τα νούμερα. Αυτό θα είχα ως παρατήρηση για τον εισηγητή, αλλά γενικά νομίζω ε, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάω Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει τον λόγο στη διαδικασία Catch the Eye. Όχι. Δίνω τον λόγο κατευθείαν στον εισηγητή. Μια που δεν βλέπω και την Κομισιόν εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ και για αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Σήμερα δεν συζητάμε ακριβώ την έκθεση, αλλά το τι κάνουμε με τις τροπολογίες. Συμφωνώ λοιπόν με αυτούς που λένε θα πρέπει να περιοριστούμε στα ζητήματα εκείνα τα οποία αφορούν την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να μην υποβάλουμε νομοθετικές προτάσεις που αγγίζουν άλλους τομείς. καμία τροπολογία δηλαδή για ζητήματα στα οποία υπάρχουν ήδη νομοθετικές πρωτοβουλίες. Δεύτερον, αναφέρθηκαν πολλά πράγματα. Χρειάζεται μια, ένας διαφοροποιημένος ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί έτσι θα έχουμε και διαφοροποιημένες δυνατότητες χρηματοδότησης. Το είπαν πολλοί συνάδελφοι και το θέμα βεβαίω νέων χρηματοδοτικών επιλογών σε σχέση με τις παλιές. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται από τη μια μέρα στην άλλη να μειωθεί δραστικά ο ρόλος των τραπεζών. Απλά θα πρέπει οι νέες πηγές χρηματοδότησης να προσθεθούν και να ενδυναμωθούν. Χρειαζόμαστε και τα δύο, και τις παλιές και τις νέες πηγές χρηματοδότησης, αλλιώς θα έχουμε χρηματοδοτικό κενό. Και τέλος, οπωσδήποτε μια τέτοια διαφοροποιημένη προσέγγιση ε, θα μπορούσε να οδηγήσει ε, μια παραπομπή στα εκτιμώντας ότι δηλαδή τα θέματα αυτά δεν είναι αντικείμενο της έκθεσης αλλά διαμορφώνουν την πολιτική άποψη. Δεν βλέπω λοιπόν κάποιο πρόβλημα εδώ, ούτε και στην ομαδοποίηση των τροπολογιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Να υπενθυμίσω πως θα ψηφίσουμε στις 13-14 ε, Ιουνίου στην Επιτροπή και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Τώρα, όπως ανακοίνωσα, πριν περάσουμε στο σημείο του Γενικού Προπολογισμού στις 6 ώρα, διακόπτω την συνεδρίαση για μερικά λεπτά. Λοιπόν, όπως είπα, επανερχόμαστε στις 6 η ώρα, σε μία ώρα. Διακόπτω τη συνεδρίαση. So, liebe. Das hatte ich auch noch nie. Okay. So, if I look around. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητέ συνάδελφοι, ή μάλλον στον ελληνικό πρέπει να το πω, γιατί στον πληθυντικό δεν έχει και πολύ νόημα. Το Έλκιν εδώ, ως επιτοπλίστων. Από το Έλκιν οι περισσότεροι. Also, sehr geehrter Berichterstatter, Κύριε Ισηγητάς, ξεκινήσουμε. 6 και 0, 2. Ξεκινάμε λοιπόν με το θέμα Γενικός Προπολογισμός τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2017. Η συγητή εδώ πέρα είναι ο Μάρκους Φέρμπερ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι είναι εδώ και ο κύριος Γιένς Γκάιερ και θα μιλήσει πρώτος. Λοιπόν, Γιένς, έχεις τον λόγο και μετά τον λόγο έχει ο ε, κύριος ε, Φέρμπερ. Κύριε Γκάιερ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφε, τρία άτομα είμαστε. Πάμε στο μπαρ εδώ πέρα να τελειώνουμε. Τι... Τέσσερα. Δεν έχουμε έρθει για την πλάκα μας. Για ούτε για να διασκεδάσουμε εδώ. Λοιπόν, να σας πω πού βρισκόμαστε. Να σας πω ποια είναι τα κέρια σημεία της διαδικασίας του προπολογισμού και πώς θα συνεχιστεί αυτή. Περιμένουμε την 25η Μαΐου, την ημέρα κατά την οποία θα ανακοινώσει η Κομισιόν τις προτάσεις της για τον προπολογισμό 2017 μέχρι τότε πέρα από τις προπαρασκευαστικές εργασίες τις κατευθυντήριες γραμμές δεν υπάρχει ποτέ άλλο να κάνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ε, προπροηγούμενη Ολομέλεια ενέκρινε τις ε, κατευθυντήριες γραμμές Δηλαδή αποφάσισαν επί της αρχής οι ομάδες πόσο επιτρέπεται να ξοδέψει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πράσινοι είναι επί της αρχής υπέρ, αλλά πήχαν γιατί δεν απορρίψαμε τον ε, ίτερ, τον αντιδραστήρα ίτερ και μας δυσκόλεψαν λίγο, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να πούμε πως οι κατευθυντήριες γραμμές είχαν την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι κατευθυντήριες γραμμές ε, τις οποίες επεξεργάστηκα εγώ και τις οποίες συμπλήρωσαν πολλοί συνάδελφοι νομίζω πως διακρίνονται από ρεαλισμό σε αντίθεση με το Συμβούλιο. Γιατί είχαμε την κατάσταση που βρήκαμε το 2016 και δεν βλέπουμε λόγο να αλλάξει, γιατί δεν έχει αλλάξει κατάσταση στον κόσμο και στην Ευρώπη. Για να πούμε ότι ο προπολογισμό του 2017 θα έχει ε, αλλάξει. Θα έχουμε παρόμοιε προκλήσει όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και τι έκανε το Συμβούλιο. Υπέβαλαν ένα έντυπο έξι ε, σελίδων. Οι τέσσερις πρώτες είναι copy-paste. Εν μεταξύ και στις τελευταίες δύο σελίδες έχουν βάλει μία παράγραφο γιατί στην αρχή νόμιζα ότι είχα τυπογραφικό λάθος μπροστά μου και ήταν το παλιό έγγραφο. Αλλά τελικά υπάρχουν κάνα δύο αλλαγές εκεί στο τέλος. Αλλά το Συμβούλιο λοιπόν δεν αντιδρά όπως εμείς να ξαναγράψει τον του 2016 κάνει κάποιες διακοσμητικές αλλαγές δηλαδή αυτό το οποίο κάνει πάντα το Συμβούλιο δίνει κάποια επαρκή ε, χρηματοδοτικά περιθώρια δηλαδή λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να αφήσει κάποιον αέρα θα έλεγα μεταξύ του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και του ανώτατου ορίου ε, του προπολογισμού για να υπάρχει περιθώριο για τα απρόβλεπτα. Οι φετινές εμπειρίες ε, και τις διαδικασίες ε, του προπολογισμού είναι ότι τα περιθώρια αυτά που παίζουν ρόλο για την εντοπίση της προσφυγικής κρίσης, δηλαδή η κατηγορία 3 εσωτερική και η κατηγορία 4 εξωτερική πολιτική, ε, εξαντλήθηκαν, έφτασαν στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Και μια που η κατάσταση δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, προφανώς τα ίδια θα γίνουν και το 17. Αυτό τουλάχιστον είναι η αφετηρία ε, με την οποία κινείται το Κοινοβούλιο. Αυτές τις κατευθύντριες γραμμές έχει υιοθετήσει και έτσι η... αυτή είναι η διαφωνία με το Συμβουλίο. Έχουμε την προσφυγική κρίση χρησιμοποιήσαμε όλα τα πολιτικά μέσα που είχαμε οτιδήποτε υπήρχε στο μεσοπρόθεσμο επίπεδο και αν δεν το κάναμε αυτό νομίζω ότι ή άλλως θα χάναμε και το παιχνίδι εντελώς οπότε ήδη έπρεπε έχουμε κάνει τον πρώτο διορθωτικό προϋπολογισμό ακριβώς για αυτό το μέσο εκτάκτου χρηματοδότησης, π.χ. για να αυξηθεί η χρηματοδότηση της Europol. Οπότε τα πράγματα ήταν περίπλοκα και θα συνεχίσουν να είναι περίπλοκα. Η οικονομική κρίση ακόμα δεν την έχουμε ξεπεράσει και αυτήν. Έχει διαφορετική ένταση και οξύτητα στα διάφορα κράτη-μέλη. Αν δεν βλέπουμε μόνο τις πρωτοπόρες χώρες, αλλά λάβουμε υπόψη τη γενική εικόνα, πρέπει να πούμε πως ε, και οι δαπάνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης αιτιολογούνται και επιτρέψατε μου είναι σαφές πως ε, το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο έτσι ως έχει αυτή τη στιγμή είναι παντός καλού καιρού όπως λέμε. Και άμα χαλάσει λίγο καιρός είναι δύσκολα τα πράγματα οπότε... θα πρέπει να ενσωματώσουμε και οτιδήποτε άλλο έχει προκύψει μέχρι το τέλος του έτους στην διαδικασία αυτή. Αλλιώς δεν γίνεται. Εγώ λοιπόν πρότεινα, α, να αναφέρω και το εξής ότι κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό και μας ενδιαφέρει ως Επιτροπή έχουμε στις γραμμές ε, του προϋπολογισμού οι οποίες το ποσό εγγύησης για το ΕΦΣΥ έχουμε 3,38 δισεκατομμύρια ευρώ αντί για τα 8 τα οποία τα θέλαμε οπότε και το να βρεθούν λεφτά για αυτή την γραμμή του προπολογισμού είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μα απασχολήσει. Λοιπόν, πρώτα στι κατευθυντήριε γραμμέ. Να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία αυτή για να δούμε κάπως ε, να συνδέσουμε αυτά τα οποία λέει η Κομισιόν για την οικονομική πολιτική με τις δαπάνες. Έχουμε τις ευρωπαϊκές οικονομικές προοπτικές, την ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη και βεβαίως το ευρωπαϊκό εξάμεινο στο οποίο γίνονται προτάσεις για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις διαρθρωτικές αδυναμίες των κρατών μελών. Και εάν καταφέρουμε ο προπολογισμό να προσαρμοστεί κάπως τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης, τότε νομίζω θα δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Βεβαίως πρέπει να ψηφιστεί κιόλας από το Κοινοβούλιο, ε. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Νεολαίας, η οποία όμως τελικά στην οποία τελικά αναγκαστικά να συμφωνήσουμε με την Κομισιόν, όχι γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι το ξεπερασμένο, αλλά γιατί η Κομισιόν λέει ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια αξιολόγηση, να δούμε τι έχει επιτευχθεί στο μέτωπο αυτό πριν ε, αφιερώσουν περισσότερα κονδύλια. Θέλουμε να συνεχίσουμε, όπως είπαμε, την καταπολέμηση της ε, φτώχειας ε, με το στόχο της στρατηγικής του ορίζοντα 2020 και να ξεκινήσουμε και με τα παιδιά. Η κατάσταση των πληρωμών έχει χαλαρώσει λίγο καθώς έχουμε νέα κονδυλία με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και η στενοπόση η οποία υπήρχε με μη εκταυμιευμένες πληρωμές έχει ξεπεραστεί και νομίζω θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ξανασυσσωρευτούν τέτοιες ε, υποχρεώσεις για να μην ξανανεύουν όπως είπαμε ε, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Και Βεβαίω, η κατάσταση όπω είπαμε κάπως ε, χαλάρωσε, δεν είναι πλέον τόσο τεταμένη, αλλά θα πρέπει το... Νομίζω το 2017 δεν θα μας δημιουργήσει ιδιαίτερου ε, πονοκεφάλους. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούμε. 25 Μαΐου θα υποβάλει την έκθεση Κομισιόν. Θα πάει στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα αλλάξει την έκθεση όπως θεωρεί αυτό σωστό. Και μετά θα έχουμε την αλλαγμένη αυτή πρόταση του ε, Συμβουλίου, στην οποία θα πρέπει να αντιδράσουμε και είμαι περίεργος να δω μετά τι θα πει η ΕΚΟΝ. Σας ευχαριστώ, Γιάννης Γκάιερ. Ο Μάρκους Φέρμπερ, ο εισηγητής μας, ε, λοιπόν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Εισηγητά, για τον προϋπολογισμό. Χαίρομαι που μετά από χρόνια έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε πάλι με αυτό το θέμα. Ήμουν επί δύο θητείες ε, τακτικό μέλος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού σε άλλες εποχές όπου δεν είχαμε μία ανάγνωση μόνο αλλά η έξυπνη ε, από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων μπόρεσαν κάπως να τα αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, Ήδη είχαμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τις κατευθυντήρες γραμμές του 2017, οπότε τα γενικά θα έλεγα τα ξέρουμε. Είμαστε σε μια αρκετά τεταμένη κατάσταση όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τις συνεννοήσεις με το Συμβούλιο. Εμείς είμαστε σε μια κάπως πιο άνετη κατάσταση εδώ πέρα. Ασχολούμαστε με κάποιες μικρές ασήμαντες γραμμές του προϋπολογισμού, αλλά το κάνουμε με την απαραίτητη σοβαρότητα. Θα ήθελα εδώ πέρα να υπενθυμίσω τις ε, τρεις ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες που έχουμε εμείς, ΕΜΠΑ, ΕΣΜΑ και ΕΙΟΠΑ, τις εποπτικές αυτές αρχές και έχουμε βεβαίως, ε, εγώ είχα ασχοληθεί και με την απαλλαγή τους και ακριβώς εκεί πέρα είδα σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας ε, το κατά πόσον είναι αναγκαία κάποια πράγματα, π.χ. υποδομές ε, που θα χρειαστεί έσμα έχουν ήδη προϋπολογιστεί για το MIFID. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει τίποτα το σοβαρό, εξάλλου βγάζουν κάθε μέρα νέες κατευθυντήριες γραμμές. Οπότε θα πρέπει να τις δούμε αυτές τις τρεις υπηρεσίες κάπως πιο λεπτομερώς γιατί όπως είπαμε αναμένουμε και την πρόταση Κομισιόν ακριβώς για τη χρηματοδότηση αυτών των ε, αποκεντρωμένων υπηρεσιών οι οποίες θα πρέπει να εργάζονται πιο αποτελεσματικά για να μην επιβαρύνουν τον καταναλωτή και τους ελεγχόμενους Μετά ε, είπαμε το τι θα γίνει γιατί θα χρηματοδοτήσουμε την οικοδόμηση δυνατοτήτων ε, για τους ε, ήταν διαφορετικά μέρη που δεν ανήκουν στο βιομηχανία. Μετά έχουμε το πρόγραμμα φυσκάλης, προπαρασκευαστικές δράσεις γιατί ήδη σήμερα το πρωί είχαμε μια συζήτηση για περισσότερη συνεργασία των φορολογικών αρχών σε σχέση με την Επιτροπή Τάξε 2 και ίσως ε, θα γίνει και μια εξεταστική επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά για τις αρμοδιότητες των φορολογικών αρχών. Οπότε θα μπορούσαμε ίσως να προετοιμάσουμε κάποιες ε, προπαρασκευαστικές δράσεις πέρα από το πλαίσιο του φυσκάλης ε, πιο εντατικά γιατί από όταν εγκρίθηκε αυτό το πρόγραμμα βεβαίως έχουν αλλάξει τα πράγματα, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε. Αυτά είναι τα τρία κορυφαία θέματα τα οποία ε, βρήκα εγώ. Έχουμε λοιπόν αφενός ε, αποτελεσματική ε, εργασία και αποτελεσματική χρήση των ε, κονδουλίων, ανταλλαγή πληροφοριών αλλά βεβαίως αυτό αφορά και την καταβολή ποσών. Μετά έχουμε αυτό το 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη χρηματοδότηση της αύξησης δυνατοτήτων των μη βιομηχανικών ενδιαφερομένων στον τομέα των υπηρεσιών με πράγματα που λέγονται Better Finance και τα σχετικά. Εγώ δεν ξέρω κανένα, καμία μήκυο η, η οποία έχει τόσα πολλά η ίδια κονδύλια. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να ακολουθεί στην πορεία που ορίζει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να βαστούν δηλαδή αυτοί στα δικά τους κονδύλια. Μετά για το Φσκάλις 2020, το ανέφερα, έχουμε ένα 7 ετές πρόγραμμα με 234 ευρώ. Ήδη δύο φορές επεξεργαστήκαμε την ε, οδηγία για τις κρατικές ενισχύσεις Οπότε ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ε, νομική βάση, αλλά θα πρέπει να δούμε το τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος φυσκάλης με κάποια άλλα συνοδευτικά μέτρα. Η γραμματεία σήμερα έστειλε ένα email και στις κοινοβουλευτικές ομάδες για κάποια προπαρασκευαστικά μέτρα για τις ανάλογες προτάσεις. Έχω κι εγώ μια ιδέα, θα τη συζητήσω με τους και οδησηγητές. Και... Βεβαίω, ε, αν κάτι από αυτά τα οποία προτείνουμε υιοθετηθεί και μπει στον ε, γενικό προϋπολογισμό, νομίζω θα είναι θετικό, αλλά για τα, τις μικρές αυτές γραμμές για τις οποίες είμαστε υπεύθυνε. νομίζω καλό είναι να ε, ληφθούν υπόψη αυτά τα οποία λέμε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Μια που οι σοσιαλδημοκράτες και το Άλντε δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, θα δώσω τον λόγο στην κυρία Σουίνμπορν για το ECR. Uh, Ευχαριστούμε τους δύο συνσύγητες. Όπως είπε ο κ. Φέρμπερ, ε, ακριβώς ήταν θέμα ε, δικό μας ε, και όσον αφορά τον προβλήμα των άλλων υπηρεσιών, οπότε θα πρέπει να δούμε, θα μην το πράγμα το πώς ήταν για τις προηγούμενες χρονιές, μιλούσαμε για την απαλλαγή και αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι δεν μπορούσαν να απορροφήσουν τα κονδυλιάρα. δεν μπορώ τώρα να εγκρίνω την αύξηση της προοικοδότησης ιδίω. Τι έκαναν το, τώρα, και με τα μέτρα δευτέρου επίπεδου, έχουν αρχίσει τώρα να μου τη δραστηριότητα, αλλά βέβαια όπως είπε ο κύριος ε, Φέρμπερ, ε, χρειάζεται να υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση για πληροφορική, ε, οπότε ας μείνει η δομή όπως έχει τώρα. Και να δούμε τι θα γίνει με ε, τη συμβολή της ε, αγοράς όπως προβλέπει το καταστατικό ε, για όσους έχουν άμεση υποπτία. Έσμα στους μηχανισμούς πιστολυπικής αξιολόγησης και λοιπά. Οπότε θα πρέπει να εξεταστεί πάντοτε η νομιμότητα των οργανισμών αυτών και να δούμε τι γίνεται με τους οργανισμούς τους εποπτικούς. Επίσης, βλέπουμε ότι τώρα οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού ελέγχουν την ίσα, αλλά παραμένει κοινωνικό χαρακτήρα αυτή. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα πρόστιμα. ίσα θα ήθελε να κρατήσει την κατάσταση όπως είναι τώρα σε σχέση με τον προπολογισμό της για τα ε, πρόστιμα. Άρα, να μην χαλάσουμε την ισορροπία που υπάρχει τώρα και να συνεχίσει η ίσα να διαχειρίζεται τα πρόστιμα και να έχουν την ευελιξία που θέλουν ότι έχουν σήμερα και στο μέλλον. Ευχαριστώ μια που δεν υπάρχουν άλλοι σκιώδεις εισηγητές. Να δώσω το λόγο στον άλλο συνάδελφο. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο σε δικασία του KTI. Ε. Όχι. Οπότε δίνω ξανά το λόγο στον κύριο Φέρμπερ. Μια που δεν υπάρχει ούτε κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να συνεδριάσουμε υπό την ηγεσία σας, μια που δεν είναι εδώ πέρα και ο πρόεδρος. Ε, ή, είμαι ο πρόεδρος, οπότε θα είμαι αναγκασμένος να δώσω τον λόγο στον εαυτό μου και δεν θα ήθελα να δώσω αυτή την εντύπωση ενός ε, σφετεριστή της Προεδρίας. Λοιπόν, και θα συμφωνήσουμε, ελπίζω να πείσουμε και κανέναν άλλον και χάρηκα γιατί ψηφίζουμε αυτή την εβδομάδα στην ε, Ολομέλεια, την Πέμπτη, την, ε, ε, την έκθεση απαλλαγή για τις τρεις εποπτικές αρχές και η Επιτροπή Ελέγχου του Περιπολογισμού νομίζω κάποια πράγματα έχει δεχτεί οπότε ήδη έχει γίνει κάποια προεργασία Είμαι σε συνεννόηση και με τους ε, τρεις ε, σκιώδεις ε, εισηγητές. Να δούμε πότε θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Και βεβαίως χαίρομαι ιδιαίτερα για την συνεργασία και με τον συνάδελφο τον σκιώδη του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Φέρμπερ. Λοιπόν, το πρόγραμμα μέχρι 13 Ιουλίου έχουμε τις ε, τροπολογίες και 19 την πρώτη παρουσίαση 19 Ιουλίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες οι τροπολογίες θα συζητηθούν 31 Αυγούστου και θα γίνει και η ψηφοφορία 2 Οκτωβρίου ε, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Καλό σας βράδυ και αύριο πρωί πρωί πάλι εδώ.